Grazie colleghi della vostra Σας ευχαριστώ συνάδελφοι γιατί ήσασταν ακριβεί στην ώρα σας. Μπορούμε να ασχοληθούμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Χωρίς άλλες εισαγωγές θα δώσω το λόγο την ε, κυρία Λοκμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες ε, ορίστηκα συντάκτρια της νομοδότησης εδώ στην ΑΦΕΤ. Αδύνατον ήταν δηλαδή να εξετάσω προσεκτικά το θέμα. Πολύ σύντομα τα βασικά. Εδώ θέλουμε καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε εάν αυτό το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκπιομηχανισμένες χώρες αποτελεί μέσο εξωτερικής πολιτικής ή πολιτικής ε, ε, εμπορίου. Η συνάδελφός μου κυρία ε, Μπέρ από τους Πράσινους στο τέλος της προηγούμενης θητείας ε, συνέταξε μια γνωμοδότηση όπου έλεγε ότι πρόκειται για μέσο εξωτερικής πολιτικής. Ε, η, έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή εγκρίθηκε από την ΑΦΕΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τώρα πρωτοβουλία και έκανε ακριβώς αυτό που πρότεινε η ΑΦΕΤ, δηλαδή το σχετικά μικρό ε, χρηματοδοτικό μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες να το μετατρέψει ώστε να ε, διατεθεί σε χώρες που δεν είναι πια αναπτυσσόμενες. Για χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία ή η Μέση Ανατολή υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, ανταλλαγών τα οποία δεν εμπίπτουν στην ε, κλασική αναπτυξιακή πολιτική. Για παράδειγμα, προγράμματα ανταλλαγών ε, ε, στην επιστήμη και στην έρευνα, όπως το Erasmus Mundus, σε θέματα μεταφορικά, πολιτικά, πολιτισμικά, για να σας αναφέρω μόνο κάποια από τα θέματα. Το χρηματοδοτικό αυτό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες αν παραμείνει στην ε, Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου, το Κοινοβούλιο θα δώσει το μήνυμα ότι κάνουμε είτε, ε, πολιτική, είτε εμπορική πολιτική είτε αναπτυξιακή πολιτική, αλλά όχι εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό σήμερα θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν ο πρόεδρος μας, κύριος Αλμπερτίνη, μπορεί να, αν μπορούμε να το αναθέσουμε, να γράψει μια ε, επιστολή στην ε, Επιτροπή Προέδρων των ε, Επιτροπών για να αναλάβουμε εμείς επί την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκάλερ, που ασχολήθηκε με το θέμα. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε η ε, συνάδελφος Λόχμπίλερ ε, στο Κοινοβούλιο. Γίνεται συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση ε, μέτρων σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες όμως δεν εμπίπτουν στην κλασική αναπτυξιακή πολιτική. Και υπήρχε αυτό το κενό στα μέσα μας ε, και γι' αυτό υπήρχε η ανάγκη να δημιουργήσουμε αυτό το ICI, ώστε να έχουμε τέτοια μέτρα μόνιμα και να μην πρέπει να τα ε, εκτελούμε ως προκατακτικά μέτρα. Ε, συμφωνώ λοιπόν απόλυτα ότι δεν πρόκειται για κλασικά μέτρα. Είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Συμφωνώ λοιπόν με τη γνωμοδότηση της ε, συναδέλφου Μπέρ που υιοθετήθηκε. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα προγραμμάτων. Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών στη Βραζιλία, για παράδειγμα. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο δεν θα μπορούσε να εμπίπτει στα DCI ή, να σας το πω στα αγγλικά, διότι δεν ξέρω πώς το λέμε στα γερμανικά, EU Visibility Public Diplomacy ε, Outreach είναι ένα πρόγραμμα για την ε, διπλωματία το οποίο ε, δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την αναπτυξιακή βοήθεια ή ε, υποστήριξη για μια ε, συμφωνία ΑΖΕΑΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφος ε, όσον αφορά επιστολή του Προέδρου μας προς την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. για να προσβάλλουμε την απόφαση να δοθεί το μέσο αυτό στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Ε, ανήκει στη δική μας Επιτροπή ε, το μέσο αυτό και θα πρέπει τουλάχιστον ε, επίσης όρις με την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου να ασχοληθούμε με το θέμα. Η παρούσα κατάσταση δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στη νομική βάση. Η Κομισιόν πρότεινε το 181α της συνθήκης Ε, με συγχωρείτε, αλλά τα αριστερά μιλάνε στο τηλέφωνο. Ε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. 181α λοιπόν, ε, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχουμε, δεν θα συναποφασίζουμε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ε, να συναποφασίσουμε. και γι' αυτό προτείνουμε το 177 και το 181α ε, κατόπιν ε, γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία μα ε, τη 27η Νοεμβρίου του 2008. Συμφωνούμε λοιπόν με τη γνωμοδότηση αυτή. την υιοθετήσαμε πριν τι εκλογέ. θα πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο κανεί θέλει να πάρει το λόγο για το ίδιο θέμα. Ή μπορώ να θεωρήσω ότι το έχουμε διεκπαιρεώσει. Δεν νομίζω ότι θέλουν άλλοι να πάρουν τον λόγο. Καταγράφω λοιπόν και συμφωνώ με αυτά που άκουσα. Συμφωνώ με τον προσανατολισμό που σκιαγραφήθηκε από τους συναδέλφους. Αν τώρα το ερώτημα είναι η αρμοδιότητα και αν αφορά μόνο την ανάπτυξη, ε, δηλαδή μεταξύ των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, προφανώς είναι εκτός θέματος. Εμείς είμαστε εκτός θέματος. Εάν όμως οι σχέσεις αυτές, οι εκθέσεις αυτές αφορούν όλες τις ε, σχέσεις μας, δηλαδή μπαίνουν μέσα σε μια προοπτική εξωτερικής πολιτικής, προφανώς είναι και δική μας αρμοδιότητα. Και θα πρέπει να συνδιαχειριστούμε το όλο πλαίσιο. Επομένως, ε, εφόσον με εξουσιοδοτείτε, θα στείλω μια επιστολή προς αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζω να ξεκινήσει η διαδικασία στο εσωτερικό της διάσκεψης των Προέδρων. Και θα δούμε τι λύση θα δοθεί. Σίγουρα θα παρακολουθήσουμε την όλη διαδικασία εκ του σύνεγγης. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε το πρώτο σημείο. Πάμε στην τροποποίηση του εργαλείου για την, του μέσου μάλλον για τη σταθερότητα. Ο κύριος Μπράτνερ είναι παρόν. Η κυρία μάλλον, διορθώνει ο πρόεδρος, θα της δώσω το λόγο για να παρουσιάσει το θέμα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Το θέμα είναι το μέσο σταθερότητας. Η συνάδελφος Αγγέλη Καμπέρα από τους Πράσινους ε, ήταν η συγγήτρια. Εγώ πρόσφατα εξελέγην, πρόσφατα άρχισα να δουλεύω πάνω στο θέμα αυτό ε, και όπως είπε η συνάδελφός μου ε, η κυρία Λόχπιλερ είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με το έγγραφο που λάβαμε από την Κομισιόν. Θα γνωρίζετε ότι πρόκειται για πρόσφατο μέσο, το μέσο σταθερότητας και η Επιτροπή πρότεινε λίγες τροποποιήσεις η μία έχει να κάνει με μία υπόθεση δικαστική. Σε τι βαθμό η Κομισιόν ε, επιτρέπεται να αποφασίζει για θέματα μικρών ε, όπλων. Ε, το δικαστήριο αποφάσισε ότι και η Κομισιόν έχει αρμοδιότητα στο θέμα αυτό, όχι μόνο το Συμβούλιο και γι' αυτό θέλει να αναγνωρίζεται αυτό στο μέσο αυτό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την απόφαση και την πρόταση της Κομισιόν. Άλλη πρόταση είναι με τη χρηματοδότηση αυτή να ε, είναι ανοιχτές προμήθειες ε, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Ε, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελβετία, αφορά και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα να διευρύνουμε την παρούσα βάση. Η το άλλο σημείο που προτείνουν είναι αύξηση για το άρθρο 4.1, ε, αύξηση ε, του ύψους 10% και από ό,τι καταλαβαίνουμε από την Επιτροπή, είναι το μέσο που είναι πιο εύκολο να δαπανηθούν τα χρήματα, διότι όσον αφορά το προσωπικό και τα προγράμματα, μπορούν να υιοθετήσουν περισσότερα Πιστεύουμε επίσης ότι είναι τομέας όπου μπορούμε να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα για να δεχτούμε την αύξηση αυτή όμως ε, θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική στρατηγική στον τομέα αυτών. Ε, πρόκειται για ε, ένα όραμα πιο μακροπρόθεσμα. Γνωρίζουμε πράγματα για λίγα από τα προγράμματα αυτά ένα κέντρο στη Μόσχα, ένα αντιτρομοκρατικό πρόγραμμα στο Αλγέρι, ένα πρόγραμμα ναρκωτικών από το Αφγανιστάν. Υπάρχουν όμως και άλλα προγράμματα εδώ, για τα οποία δεν γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Η γραμματεία του Κοινοβουλίου προσπάθησε να λάβει πληροφορίες, ιδιαίτερα σχετικά με το κέντρο στο Αλγέρι. Εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί, αλλά δεν έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα αυτό. Αντιτρομοκρατικό κέντρο στο Αλγέρι είναι κάπως ευρία έννοια. Θα θέλαμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό, προτού να συμφωνήσουμε στην αύξηση του προπολογισμού, στον, της γραμμής του προπολογισμού για τον τομέα αυτών. Δύο ακόμα παρατηρήσεις. Το πρώτο το ανέφερα ήδη, σχετίζεται με το κέντρο στο Αλγέρι. Θα θέλαμε να ε, υποβάλλονται εκθέσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν αρκετέ αξιολογήσει που δεν έχουμε λάβει, που τι έχει λάβει το Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρόσβαση στι εκθέσει αυτέ. Το άλλο θέμα είναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα ε, τελική σχέση οικοδόμησης της ειρήνης και θα θέλαμε πολύ να δούμε την στρατηγική της Επιτροπής, διότι μέχρι τώρα είχαμε διασκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια, αλλά δεν έχει γίνει η πραγματική δουλειά επί της ουσίας. Θα θέλαμε μια σαφή προοπτική της Κομισιόν σχετικά με το τι σκοπεύει να κάνει μέσα στον επόμενο χρόνο. Θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, διότι είναι σημαντικό για μας και δεν βλέπουμε να έχει εφαρμοστεί ακόμα σωστά. Και τελευταία παρατήρηση, Δυστυχώς, ε, λόγω πολιτικού συμβιβασμού, μεγάλο μέρος ε, του μέσου σταθερότητας έχει χρησιμοποιηθεί για ε, το μέσο για τα τρόφιμα. Είχε προταθεί αρχικά να πάρουν, να παρθούν χρήματα και από τον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Ε, μέρος του μέσου σταθερότητας ε, θα πρέπει να ε, το αφήνουμε στην άκρη για περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης και γι' αυτό δεν θέλουμε να προγραμματίσουμε όλη τη διάσταση των πόρων από την αρχή, αλλά δεν θα είναι απλά ένα γενικό απόθεμα το μέσο αυτό. Δεν μπορούμε απλά να το χρησιμοποιούμε όποτε μας βολεύει για ε, προγράμματα που θα πρέπει να ε, χρηματοδοτηθούν από άλλα μέσα όπως είναι το θέμα των τροφίμων. Θα θέλαμε να το συζητήσει αυτό και η Επιτροπή του Προϋπολογισμού, διότι έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός κατά 20% εξαιτίας αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Μίλλερ για να μας εξηγήσει γιατί η Κομισιόν ζήτησε αυτή την πρόταση τροποποίησης. Γιατί την έκανε μάλλον αυτή την πρόταση τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Έχετε το λόγο κύριε Μίλλερ. Να πω δύο αρχικά λόγια εισαγωγικά για την ενδιάμεση αναθεώρηση των μέσων ε, εξωτερικών σχέσεων. Καταρχάς του μέσου σταθερότητας. Η πρόταση είναι τμήμα ε, ενό πακέτου προτάσεων που έχουμε υποβάλει. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα συμπεράσματά μας για τη γενική κατάσταση των μέσων είναι ότι δουλεύουν καλά, ότι μας έχουν δώσει μια επαρκή βάση για την εξωτερική πολιτική. Δεν έχουμε ουσιαστικέ δυσκολίε στην εφαρμογή κανενός από τα μέσα. Και αυτό φαίνεται ε, στο γεγονός ότι το ύψος της βοήθειά μας έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Τα βασικά πορίσματα της ε, έκθεσης είναι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που δεν ε, θεωρούνται ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και προτείναμε να το επιλύσουμε ε, στο πλαίσιο των μέσων των εκβιομηχανοποιημένων χωρών. Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συζητήσουμε εμεί ω Κομισιόν τα εσωτερικά σας του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν είσαστε αρμόδια, μια άλλη επιτροπή. Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε την ενδιάμεση έκθεση ως πακέτο και οποιοδήποτε μέτρο που θα προωθήσει το Συμβούλιο, ε, το, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο για να έχουμε μία εξισορροπημένη πολιτική θα μας βοηθούσε. δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κανένα ε, πρόγραμμα ε, υπό το μέσο των εκβιομηχανοποιημένων χωρών ε, μέχρι τον Ιανουάριο, αν δεν έχουμε όλες τις προτάσεις μέχρι τον Ιανουάριο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα και πρέπει η χρηματοδότηση να συνεχιστεί. Το είπαν και κάποιοι βουλευτές ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα προς το συμφέρον τη κοινότητα που έχουν να κάνουν με οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία με τρίτες χώρες. Επίσης, θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και το ευρωπαϊκό τμήμα του Erasmus Mundus, να στείλουμε καθηγητές και φοιτητές στο εξωτερικό. Από κάπου πρέπει να το πληρώσουμε αυτό. Και νομίζουμε ότι πρέπει να πληρωθεί αυτό από το μέσο για τις εκβιομηχανοποιημένες χώρες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα διακυβευθούν. Δεν θα μπορέσουμε να ξοδέψουμε το προϋπολογισμό αν δεν υλοποιηθούν, θα εγκριθούν αυτά τα μέτρα έγκαιρα. Νομίζω ότι υπάρχει η φιλοδοξία σε εσά και στο Συμβούλιο να υπάρξει συμφωνία μέχρι το, μέλος, μέχρι το τέλος του χρόνου και ελπίζω λοιπόν να μας υποστηρίξετε στην προσπάθειά μας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση που έχουμε τώρα μπροστά μας για το μέσο σταθερότητας, ο κύριος Μπράτνερ, ο εισηγητής, ε, συνόψε την πρόταση πολύ σωστά. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλα τα θέματα που έχετε θέσει. Ε, η κυρία Μπάρτνα, διορθώνει ο μιλητή, θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει κάποιε από τι πληροφορίε. Θα το κοιτάξω με του συναδέλφου και θα κοιτάξω γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Και θα δω αν μπορούμε τώρα να σα δώσουμε τι πληροφορίε και μάλιστα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Κατέγραψε επίση τα σχόλια για την εταιρική σχέση με σκοπό την οικοδόμηση της ειρήνης. Οι αρμόδιοι συνάδελφοί μου δεν είναι εδώ ακόμα. Ίσως όταν φτάσουν, καλό θα ήταν να τους δώσετε τον λόγο. Τώρα δίνουμε, αυτή τη στιγμή υπογράφουμε τα, τις συμβάσεις για τα πρώτα δάνεια Ξέρω ότι οι συνάδελφοι τώρα σκέφτονται τις επόμενες φάσεις. Θα το αφήσω το θέμα αυτό όταν φτάσουν να το παρουσιάσουν οι ίδιοι. Αυτό που είπε η κυρία Μπάρτνερ για τον προϋπολογισμό για του μέσου σταθερότητα είναι σωστό. Αλλά αυτό είναι θέμα της Επιτροπής, νομίζω, προπολογισμών του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται εκεί, δυστυχώς. Πρόεδρε, η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει τους βουλευτές για οποιαδήποτε ερωτήματα έχουν σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση έκθεση συνολικά και τα μέσα για τα οποία η Επιτροπή σας είναι αρμόδια. Μπορούν να αποτανθούν σε μένα και εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Όταν έρθει ο αρμόδιος συνάδελφός σας θα επανέλθουμε στο σημείο. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να σας δώσω ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα λάβετε το τελικό προσχέδιο της έκθεσης και στις 20 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία για την παρουσίαση των ε, τροπολογιών. Εκτιμούμε ότι μέχρι τις 4-5 Νοεμβρίου η συζήτηση για την ε, έκθεση και για τις τροπολογίες θα γίνει, ούτως ώστε να πάμε μετά στις 10 Νοεμβρίου σε ψηφοφορίες. Και με συναπόφαση ένα μήνα μετά 14-15 Δεκεμβρίου να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. μου είπαν ότι δεν είναι παρούσα η κυρία Λάτφορντ, η συγγήτρια για το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη. Σταματάω λοιπόν την συνεδρίαση, κάνω ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών, περιμένοντας την συγγήτρια. Ούτως ή άλλως έχουμε διεκπαιρεώσει πολύ γρήγορα τα προηγούμενα σημεία και ίσως δεν αφήσαμε αρκετό χρόνο στη συνάδελφο να φτάσει εγκαίρως. Σταματάω λοιπόν μόνο για πέντε λεφτά. Bene, eh, mi viene, eh, mi viene comunicato in questo momento... Μόλις μου κοινοποίησαν ότι η συγγήτρια, η κυρία Λάτφορντ, έφτασε. Επομένως, μπορούμε να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ζητώ συγγνώμη. Un attimo di attenzione ai colleghi. Eh, sedetevi per favore. Παρακαλώ συνάδελφοι, καθίστε για να ξεκινήσει η συζήτηση. Πρόκειται για τον κατάλογο τρίτων χωρών, οι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Θα μιλήσουμε επίσης και για τους υπηκόους χωρών, των οποίων οι υπήκοοι δεν υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την πρόταση της Κομισιόν που κατήργησε την υποχρέωση αυτή για την πρώην ε, Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας, ε, για τη Σερβία και για το Μαυροβούνιο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λάτφορντ για να μας παρουσιάσει το σημείο αυτό. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ε, λυπάμαι αν σας καθυστέρησα λιγάκι γιατί μόλις έφτασα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να τονίσω τα σημεία που απασχολούν αυτή την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο γενικότερα. Διότι εμείς υποστηρίξαμε την ελευθέρωση υποχρέωσης θεώρησης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων κάτι το οποίο εντάσσεται στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης και βεβαίως αυτές οι χώρες θα είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που πληρούνται τα κριτήρια και οι διαδικασίες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αν το έχετε λησμονήσει, ότι στις ε, χώρες της πρώην Ιουκοσλαβίας οι πολίτες μπορούσαν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Άρα, οι χώρες που υπόκεινται σε θεώρηση, ε, αυτό ακριβώς αποτελεί μία παλινοδία σε σχέση με ό,τι συνέβαινε αρκετά χρόνια πριν. Δεν χρειάζεται να απαριθμίσω τους λόγους, γιατί είναι σημαντική η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τις επαφές μας, και για τον γενικότερο διάλογο, τη διάδραση, η οποία θα βοηθήσει αυτές τις χώρες να εξοικειωθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατανοήσουν τα πλαίσια συνεργασίας και να προετοιμαστούν για μια ενδεχόμενη ένταξη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ευπρόσδεκτη και ο Επίτροπος Ρεν πρόσφατα ήρθε ενώπιον της Επιτροπής μας μετά από πρόσκληση και μας εξέφεσε το ζήτημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προβάλλουμε ορισμένες εγγυήσεις έτσι ώστε να επιτευχθούν ορισμένες ε, προδιαγραφές ως προς την, ε, τον οδικό χάρτη ελευθέρωσης των ε, θεωρήσεων. Δηλαδή χρειάζεται μια ευρύτερη, γενικότερη ε, όθηση, όπως ισχύει στην ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, όπου είμαι συνεισηγήτρια μαζί με την κυρία Τάιον. Θα πρέπει λοιπόν να εντάξουμε αυτές τις πέντε χώρες στα ίδια πλαίσια, διότι υφίσταται ο εξής κίνδυνος. Μπορούμε να λάβουμε τη Βοσνία Ερσεγοβίνη και την Αλβανία και να τις ξεχωρίσουμε, να τις απομακρύνουμε από αυτή την απόφαση και να πούμε ότι το 2010 θα γίνει μια διασάφηση, δηλαδή να υπάρξει μια καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Προτείνω λοιπόν εδώ, σε σχέση με τις πέντε χώρες, αυτό προτείνω είναι το εξής να κρατήσουμε την βασική ιδέα ότι η Σερβία και το Μαυροβούνιο πληρούν τους όρους μέχρι ότου εγκριθεί ο παρόν κανονισμός, κάτι το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι η Σερβία μας ανέφερε ότι θεωρεί ότι πληρεί τους όρους, αυτό δεν το σχολίασε βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είπαμε ότι σε σχέση με την ε, Αλβανία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ότι η εξαίρεση από το καθεστώς θεωρήσαν θα ισχύσει χωρίς χρονοτριβή μόνο όταν οι χώρες αυτές ε, πληρούν τους όρους που ορίζονται στον οδικό χάρτη και όταν αυτή η αξιολόγηση δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα των κοινοτήτων. Δηλαδή, τις κρατάμε στην ίδια νομική διάρθρωση του κανονισμού, αλλά η εφαρμογή κάθε αυτή της ελευθέρωσης από το καθεστώς θεωρήσεων θα βασίζεται σε μια αξιολόγηση από την Επιτροπή ότι τηρούνται δηλαδή οι προδιαγραφές. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διενεργείται μηνιαίως και θα κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο καθώς και τις ενδιαφερόμενες χώρες. Αυτό ε, δεν ε, το είδαμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα το ζητήσω από, την, από τον εισηγητή, διότι πρόκειται για μια συνεχή αξιολόγηση έτσι ώστε αυτές οι χώρες να βρίσκονται σε γρήγορση και εμείς ως ε, θεσμικά όργανα να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες για να πληρούν τους όρους αυτούς. Ως προς το κοσυφοπέδιο, και ασχολούμαι τώρα με, πριν ασχολήθηκα με τροπολογία 2, τώρα με την 1, το κάνω αντίστροφα δηλαδή, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει με το διάλογο απελευθέρωσης θεωρήσεων και να καταρτήσει οδικό χάρτη για το κοσφοπέδιο, όπως ισχύει με τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ε, υπό την επιφύλαξη του κατά πόσο αναγνωρίζουμε το κοσυφοπέδιο ως ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι 22 κράτη ε, έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπέδιο ενώ 5 δεν το έχουν αναγνωρίσει, θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα του κοσυφοπεδίου έτσι ώστε να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες χώρες χωρίς χρονοτριβή. Και βεβαίως ε, υπάρχουν πρακτικοί λόγοι γιατί ακριβώς θέλουμε όλοι να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Για να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στην ε, εφαρμογή του καθεστώτος περί υπηκότητας μιας γειτονικής χώρας. Εάν δηλαδή μερικές χώρες ε, δεν υπόκεινται σε αυτό το καθεστώς, ενώ άλλες υπόκεινται στο καθεστώς των θεωρήσεων. Δεν θέλουμε βεβαίως να το παίξουμε κασάνδρες και να θεωρήσουμε ότι ορισμένες χώρες μεταβαίνουν σε μία, μία χώρα, μάλλον υπήκοοι μίας χώρας μεταβαίνουν σε μία γειτονική, γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν ίσοι και δίκαιοι όροι πρόσβασης. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ένα καθεστώς ε, επαληθεύσεων. Βεβαίως κανένας μας δεν το επιθυμεί αυτό. Πρέπει να ασκηθεί πίεση σε ορισμένες εμπλεκόμενες κυβερνήσεις, δηλαδή ότι θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος στις χώρες οι οποίες δεν πληρούν απολύτως τα, τις οριοθετήσεις αυτές. Και εάν η Επιτροπή έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία μέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης, μπορούμε να ζητήσουμε και μία μηνιαία αξιολόγηση όπως ζήτησα από την, βασική, από την κύρια εισηγήτρια, νομίζω ότι έτσι θα, ε, θα έχουμε μια εποπτεία και θα ασκήσουμε και πίεση, πολιτική πίεση σε αυτές τις χώρες, διότι οι υπήκοοι της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας θα δουν ότι ο δρόμος απελευθέρωσης από το καθεστώς των θεωρήσεων βρίσκεται στα χέρια της δικής τους κυβέρνησης και δεν χρειάζεται, δεν, δεν χρειάζεται να μείνουν πίσω από το πρώτο κύμα χωρών. Και πρόθεση μου είναι, και ελπίζω να με υποστηρίξετε, είναι να μικρύνει το χάσμα ως προς τον αριθμό μηνών μεταξύ των πρώτων χώρων που θα ακολουθήσουν την ελευθέρωση και το δεύτερο κύμα που θα είναι η ε, Αλβανία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη και ελπίζουμε και το Κωσυφοπέδιο να μην έχει μείνει πολύ πίσω για όλα τα ευεργετήματα, για όλους τους λόγους τους οποίους σας προανέφερα. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που δεν πρόφερα καλά το όνομά σας. Λάτφορτ λέγεστε. Ε, είχα κάνει λάθος και για την υπηκότητά σας. Μουνίθ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, αλλά και ένα συγκεκριμένο τεχνικό περιεχόμενο. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά θέματα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας που δεν πληρούν τους όρους απελευθέρωσης θεωρήσεων, αλλά η λύση της εισηγήτριας είναι να δούμε πώς μπορούν να μπουν στις διαπραγματεύσεις και πότε πληρούν τους όρους έτσι ώστε να ισχύσει αυτή η πολιτική. Αυτό είναι ένας πολύ καλός συμβιβασμός για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Αλλά για το κοσυφοπαίδιο το θέμα είναι περίπλοκο, γιατί θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με διαπραγματεύσεις για να μιλήσουμε για έναν οδικό χάρτη για την απαλλαγή από το καθεστώς ε, θεωρήσεων, για την επανειστοχή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να αναφέρουμε στην τροπολογία ότι με την επιφύλαξη όλων των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό είναι απαράβατος όρος. Θα πρέπει λοιπόν, αν αναφερθούμε στο κοσυφοπέδιο, θα πρέπει να μιλήσουμε για το καθεστώς του κοσυφοπεδί και με βάση το ψήφισμα 1244 των Ηνωμένων Εθνών υπό την επιφύλαξη αυτή. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση. Και γι' αυτό νομίζω ότι η τροπολογία 3 της ε, έκθεσης της Τάνια Φαζών στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μπορεί να γίνει αποδεκτή, γίνεται περισσότερο αποδεκτή όταν λέει υπό την επιφύλαξη του στάτους του Κωσίφου πεδίου, σύμφωνα, και εγώ θα ήθελα να προσθέσουμε, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αυτό έτσι δηλαδή η τροπολογία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από εμάς. Αν αναφερθεί και το εν λόγω ψήφισμα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μόνιχ, η συνάδελφος Λούνατσεκ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους συντάκτες της νομοδότησης ε, για την νομοδότηση αυτή που προτείνει και κάποιες τροπολογίες. Εκτιμώ την... το σχέδιο πρότασης που είχαμε από την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και την ε, πρόταση της ΑΦΕΤΕ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κοινό όραμα, ένα κοινό πακέτο για όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευ... Ευρώπης. Όπως ε, έχει πει η Βαρόνι Λάτφορντ στο παρελθόν, ε, πριν 20 χρόνια ο κόσμος μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα από τις χώρες της πρώην Ιουκοσλαβίας σχεδόν σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι νέοι τώρα που ξέρουν ότι οι γονείς τους μπορούσαν να το κάνουν αυτό, δεν έχουν αυτές τις ελευθερίες. Ξέρουμε ότι ο εθνικισμός και ο εξτρεμισμός αποτελούν ε, πρόβλημα στις χώρες αυτές. Το να ταξιδεύουν λοιπόν, ιδιαίτερα οι νέοι σε άλλες χώρες, ε, να γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς, ε, θα το έχετε νιώσει κι εσείς. Είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ για να μάθει κανείς ε, να δέχεται τους άλλους, να δέχεται τις θέσεις των άλλων, ε, να δέχεται την ποικιλομορφία, να δέχεται τις απόψεις των άλλων ακόμα και αν δεν τις συμμερίζεται. Η ιδέα λοιπόν του να συμπεριλάβουμε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον κανονισμό αυτό ε, είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Το εκτιμά και η ομάδα μου όσον αφορά τις λεπτομέρειες στο κείμενο. Εκτιμώ αυτό που υπόθηκε ότι η Αλβανία και η Βοσνία Ζεγοβίνη ε, συμπεριλαμβάνονται στην ε, τροπολογία με το κείμενο που προτείνεται. Όσον αφορά το κοσυφοπαίδιο, ε, δέχομαι το κείμενο που προτείνει η κυρία Λάτφορτ, διότι και εγώ έχω πάει στο Κωσυφοπαίδιο. Βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κωσυφοπαίδιο. Ε, συνομίλησα με πάρα πολλού ανθρώπου και έχω μια σαφή εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε στους πολίτες του Κωσυφοπεδίου μια προοπτική. Προοπτική ότι θα συμμετάσχουν και εκείνοι στο πακέτο αυτό, θα μπορούν και εκείνοι να ταξιδεύουν. Στην ε, Πρίστινα από τον Υπουργό Εσωτερικών ε, ε, έλαβα την εντύπωση, μάλλον μου είπε ρητά, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει έναν οδικό χάρτη με σαφείς ιδέες σχετικά με το πόσο μπορούν να ε, πληρωθούν όλα τα κριτήρια που ισχύουν και για τις άλλες χώρες. Εκτιμώ λοιπόν ιδιαίτερα το κείμενο όπως προτάθηκε με την τροπολογία. Όπως είπε ε, η συντάκτη, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει μήνυμα σαφές ότι, ότι πρόκειται για τρόπο που ισχύει για όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας αυτής, δεν ισχύει μόνο για μερικούς. Θα είναι πρόβλημα εάν μία ή δύο χώρες δεν έχουν την ίδια προοπτική, διότι τότε οι πολίτες τους θα προσπαθούν να λάβουν υπηκότητα κάποιας γειτονικής χώρας. Θέλουμε όμως και εμείς να γνωρίζουμε ποιο είναι ο πολίτης ποιας χώρας ε, στη χώρα, στην περιοχή αυτή, στην περιφέρεια αυτή. Όσον αφορά τις ε, ανησυχίες ε, της Ισπανής συναδέλφου, ναι, γνωρίζουμε ότι δεν έχουν αναγνωρίσει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κωσυφοπαίδιο. Αλλά και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου χώρες που δεν έχουν αναγνωριστεί από όλους έχουν ότι και για τέτοιες χώρες έχουν υπάρξει ε, τέτοια καθεστώτα, όπως ε, το Ταϊβάν. Θα είναι καλό για τους ανθρώπους του κοσφοπεδίου, ας μην μιλήσουμε για το καθεστώς, για τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους νέους, θα είναι σημαντικό να έχουν την προοπτική ότι θα συμμετέχουν στην Ευρώπη. Ανήκουν στην Ήπειρο αυτή και έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ένα αίτημα έχω αν ε, συμφωνεί η συντάκτρια. Θα μπορούσα να τους περιλάβουμε στην αιτιολογική έκθεση στην αρχή. Όπως ε, σας ε, είπα ήδη, η κυβέρνηση του Κωσοφοπεδίου ετοιμάζει ο χάρτη. Εάν συμφωνείτε, θα μπορώ να το, να το υποβάλω και ως τροπολογία φυσικά, θα πρότεινα λοιπόν ε, στην, ε, στην αρχή, στα να πούμε ότι ε, επικροτούμε την προσπάθεια των αρχών του Κοσφοπεδίου να υιοθετήσουν οδικό χάρτη. Και μία ερώτηση έχω ειδικά προς την Κομισιόν και ένα αίτημα. Το θέμα των... της φύλαξης των συνόρων ανάμεσα στη Σερβία και στο Κοσφοπέδιο νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ε, προς τη Σερβία ότι θα πρέπει να ισχύει να ισχύουν οι ίδιοι έλεγχοι στα σύνορα αυτά με οποιοδήποτε άλλο διεθνώ αναγνωρισμένο σύνορο, διότι αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα ελέγχου της κυκλοφορία ε, και των ανθρώπων που ε, θα περνούν τα σύνορα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι ένα αίτημα προς την Κομισιόν. Δεν ξέρω αν θεωρείτε δεν, δεν ξέρω αν πρόκειται να ζητήσετε αυτό το πράγμα από τη Σερβία. Δηλαδή, ο έλεγχο που θα ισχύει στο σύνορο αυτό να είναι ο ίδιο που ισχύει ε, σε όλα τα άλλα διεθνή σύνορα. Επίση, μια διευκρίνηση για όσου από εσά μπορεί να διαβάσατε ε, άρθρο του BBC για την επίσκεψή μου στο Κοσμοπέδι την προηγούμενη εβδομάδα, όπου αναφέρεται ότι λέω ότι ε, εμεί η αποστολή προ την νοτιοανατολική Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα φροντίσουμε ε, οι χώρες ε, που ε, δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο θα θα φροντίσουμε να αναγνωρίσουν το κοσφοπέδιο. Να κατεστήσω σαφέ. Δεν μιλούσα εκ μέρου ε, τη αποστολή, μιλούσα εκ μέρου του κόμματος, τη πολιτική μου Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συμφωνήσω με την συνάδελφο Λούνατσεκ. Θα ήθελα να τονίσω τη θέση αυτή. Καταρχήν, θα πρέπει να είναι σαφές ότι όλοι, και ιδιαίτερα στη Γερμανία και στην Αυστρία, έχουμε ζήσει στη δεκαετία του 70 ε, τους ανθρώπους της Ιουγκοσλαβίας ε, που ταξιδεύαν ελεύθερα ενώ τώρα είναι απομονωμένοι στη χώρα τους. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σκεφτούμε πολιτικά εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. <clears throat> Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραβλέψουμε τα τεχνικά ε, προβλήματα και προβλήματα ασφαλείας, αλλά είναι πολιτικό θέμα, γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω τη θέση της ε, συναδέλφου Λάτφορντ. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι και για λόγους ασφαλείας η συνάδελφος Λάτφορτ ε, και εγώ συμμετείχαμε επί 10 χρόνια στην ε, ίδια επιτροπή και δεν ε, υποτιμούμε τα θέματα ασφαλείας, αλλά δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τη σταθεροποίηση των χώρων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οποιαδήποτε ε, έλλειψη σταθερότητας ε, θα επηρεάσει εμάς και την ε, κατάσταση ασφαλείας μας. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε ε, και τους πολίτες της της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στην Μακεδονία, όπου υπήρχε τα τελευταία χρόνια μια διαδικασία όπου όσοι μπορούσαν ζητούσαν βουλγαρική υπηκότητα λόγω του καθεστώτος για τις θεωρήσεις και αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Εάν λοιπόν φανταστούμε το, ίδιο ε, για την Βοσνία-Ζεγοβίνη, αυτό μπορεί να αποτελέσει το τέλος του κράτους αυτού. Είναι λοιπόν καυτό το θέμα και όσον αφορά την ασφάλεια. Και τρίτο και τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι το κοσμοπέδιο. είμαι σκιώδης εισηγητής εδώ και πέντε χρόνια ε, για το κοσφοπέδιο και μπορώ να σας πω ότι οι συνάδελφοί μας από χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο Ε, δεν σημαίνει ότι μπορούν να επιβάλλουν τη θέση τους ε, στην πλειοψηφία ε, των ε, των ε, ε, κρατών μελών. Με 75% ε, τα 100 πλειοψηφία έχουμε υιοθετήσει έκθεση στην οποία λέμε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάμε την αναγνώριση του κοσμοπεδίου. Έχουμε ζητήσει πολύ σαφώς την αναγνώριση αυτή. 20 από 25 κράτη-μέλη έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο και πιστεύω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να συμφωνήσουμε να γίνονται η ε, μειοψηφία να, να γνωρίζει τη θέση της πλειοψηφίας ε, και να την ε, σέβεται και όχι να προσπαθεί να επιβάλλει τη θέση της. Ε, δεν υπάρχει εδώ η αρχή της ομοφωνίας. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει ποιον θέλει να γνωρίσει. 22 κράτη-μέλη έχουν ε, υιοθετήσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, το, οι άνθρωποι του κοσμοπεδίου έχουν υποφέρει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ε, στα Βαλκάνια. Ε, δεν υπάρχει ομοφωνία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι νέοι εκεί εξαρτώνται από τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Ευρώπη. Και θα ήταν περίεργο να παρεμβαίνουμε εκεί με πολλά χρήματα να ανοικοδομούμε τη χώρα να μιλάμε για ευρωπαϊκά πρότυπα ενώ ταυτόχρονα να ε, αποκλείουμε τους ανθρώπους αυτούς, ε, να τους απομονώνουμε ε, στη, μικρή αυτή περιοχή. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με τη συνάδελφο Λάτφορντ και θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι όποιος πληρεί τα κριτήρια μπορεί να συμμετέχει εκτός από το κοσφοπέδιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Προβέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα-δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω. Η συνθήκη προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη γνώμη του στα πλαίσια μιας διαβούλευσης για τις προτάσεις της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Η συγγήτρια τώρα προτείνει ότι για δύο χώρες το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρετηθεί από τα προνόμια του και να αφήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει. Αποφασίσει δηλαδή για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε τις ε, εξαιρέσεις. Ή θα θεωρήσουμε ότι η συνθήκη ισχύει και ότι είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να ισχύει για τα πάντα και για όλους αν, όπως προβλέπει η συνθήκη, τα όσα προβλέπει η συνθήκη δεν θεωρούνται επίκαιρα και κατάλληλα, θα πρέπει να την αλλάξουμε. Αυτός ο δικός χάρτης δεν προβλέπεται ως διακριτική μεταχείριση εναντίον κάποιων χωρών. Προβλέπει κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου, την ε, διοικητική σοβαρότητα και την ασφάλεια στις χώρες που υποδέχονται άτομα τα οποία διέρχονται τα σύνορα. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν προβλήματα τρομοκρατίας και εγκληματικότητας που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτές οι παράμετροι, αυτή η τεχνική ας πούμε πορεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί διάκριση εναντίον κάποιων. Επίσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για διακρίσεις αν υπάρχει έλλειψη προϋποθέσεων, αν δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει πρώτα να πληρωθούν προκειμένου να καταργήσουμε την υποχρέωση θεωρήσεων. Εγώ λοιπόν μετά από αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν ως έχει. Σας ευχαριστώ κύριε Προβέρα και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τάλερ. Ε, ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό προς την κυρία Λάτφορ, την εισηγήτριά μας, γιατί νομίζω ότι έκανε μια θαυμάσια δουλειά και υποστηρίζω την κατεύθυνση που μας και αγράφησε. Επίσης πιστεύω ότι το σχέδιο έκθεσης της ε, κυρίας Φαγιών, της ε, Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, είναι καλό έγγραφο και επίσης θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Τώρα, θα ήθελα να τσεκάρω κάτι, να μου πει κάτι η Κομισιόν. Το πώς έχουν ληφθεί αποφάσεις δηλαδή τους τελευταίους μήνες, τέσσερις-πέντε μήνες. Όλοι γνωρίζουμε ότι στις αρχές Ιουλίου, όταν η Κομισιόν πρότεινε να δοθεί αυτό το καθεστώς ε, για την Σερβία, Μαυροβούνιο και Φιρόμ χωρίς την υποχρέωση θεωρήσεων, τροποποιώντας τον κανονισμό του Συμβουλίου, μόνο η Φιρόμ εκείνη την εποχή πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις του οδικού χάρτη που είχε θεσπίσει η ίδια η Κομισιόν. Επίσης γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν αποφάσισε να προσθέσει στην λευκή, στο λευκό κατάλογο τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, χωρίς να πληρούν όμως τις προϋποθέσεις αυτών των οροσίμων, τα ορόσημα τα οποία είχε καθιερώσει η ίδια η Κομισιόν. Η Βοσνία, Ζεγοβίνη και η Αλβανία επίσης δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και κατά συνέπεια δεν έχουν προσθεθεί στην πρόταση της Κομισιόν της 15ης Ιουλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά την Βοσνία Ερζεγοβίνη, η πρόταση της Κομισιόν έλαβε κάποιες κριτικές από τα, τις χώρες της περιοχής, ε, οι οποίες είπαν ότι θα περιπλέξει την ε, διαδικασία στην περιοχή. Το ερώτημά μου είναι, η Κομισιόν πώς αποφάσισε να συμπεριλάβει κάποιες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στην πρόταση της 15ης Ιουλίου και να αποκλείσει κάποιες άλλες. Είναι σημαντικό πολιτικό θέμα. Είναι σημαντικό θέμα όταν λέμε ότι τα κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται. Ναι, συμφωνώ. Αλλά τότε θα πρέπει να τα πληρούν όλες οι χώρες. Εδώ όμως είχαμε κάποιες εξαιρέσεις. Παραδείγματος χάρη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια. Παρ' όλα αυτά συμπεριλήφθησαν στην πρόταση. Και είχαμε τη Βοσνία και την Αλβανία που δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα κριτήρια και δεν συμπεριλήφθησαν. Πώς ελήφθη λοιπόν η απόφαση. Γιατί η Αλβανία και η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν έλαβαν τις ίδιες ε, ευκαιρίες για να, δουν, να εξηγήσουν τι πρόοδο έχουν σημειώσει μέχρι το Δεκέμβριο, ας πούμε, φέτος. Ενώ κάτι τέτοιο έχουν ευκαιρία να το κάνουν η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Είναι μια απλή ερώτηση. Γιατί δεν δόθηκε η δυνατότητα σε αυτές τις χώρες γιατί στην Αντίγουα, στην Παχάμα, στο Μπαρμπέιντος, ε, στην Αντίγουα, στις Αιχέλες, Έχω, τις έχουμε αυτές προσθέσει στις χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται θεώρηση. Νομίζω ότι οι προτάσεις μας και οι προθέσεις μας και η στάση που προτείνει η κυρία Λάτφορντ ουσιαστικά διορθώνουν αυτό το πολιτικό λάθος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην δημιουργούμε επιπλέον ρογμές στα Βαλκάνια. Η Κομισιόν θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποιες τεχνικές αποφάσεις, έτσι ονομάζονται, έχουν τεράστιες πολιτικές συνέπειες μερικές φορές, όπως αυτή την περίπτωση. Προτείνω λοιπόν καταρχάς να μας απαντήσει η Κομισιόν, γιατί προφανώς ελήφθη μια πολιτική απόφαση Κάποιου να τους συμπεριλάβουμε παρότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια και να αποκλείσουμε κάποιου άλλους που επίσης δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Και συμφωνώ με την πρόταση που μας και αγράφησε η συγγήτριά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τάλερ. Και τώρα το λόγο η κυρία Πακ που είναι η συγγήτρια για τη Βοσνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με ε, τις προτάσεις της συναδερφού ε, Λάτφορτ. Μόλις γύρισα από τη Βοσνία και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια, ωστόσο όμως οι τεχνικές προϋποθέσεις εκτός από τα βιομετρικά διαβατήρια ε, πληρούνται. Γι' αυτό μπορώ να συμφωνήσω με την συνάδελφο. Γιατί εδώ δεν γράφει ε, όπως ακριβώς ε, και το, ε, για το... Γιατί δεν έχουμε εδώ το Κοσμοπέδιο και την Αλβανία όπως έχουμε για παράδειγμα το Μαυροβούνιο, διότι, διότι και εκεί δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια. Θα πρέπει να ε, δεχτούμε όλοι αυτό που γράφει η κυρία Λάτσφορτ και όσον αφορά το κοσμοπέδιο συμφωνώ απόλυτα, δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Ε, ανήκει και αυτό στη διαδικασία της Θεσσαλονίκη ε, και εάν θέλουμε να παραμείνει η ειρήνη στο κοσμοπέδιο θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε το κοσμοπέδιο να πληρεί τα κριτήρια που θα πρέπει να πετύσουμε. Δεν είμαι κατά των benchmarks, αλλά Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι και γι' αυτό πιστεύω ότι η κυρία Λάτφορτ πολύ σωστά έκανε, πολύ σωστές είναι οι τροπολογίες της και συμφωνώ απόλυτα. Όλα η κολέγα Τάν. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να πω, λέει ο κύριος ε, Τάνοκ, ότι είμαι υπέρ της ελευθέρωσης για την Σερβία ε, Βοσνία Ερσεχοβίνη και ε, Μαυροβούνιο. Ως προς το Μαυροβούνιο θα ήθελα να πω ότι στην Ποτγκορίτσα θα διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω και η Σερβία και η Μακεδονία να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς. Θα ήθελα να ότι διαφωνώ με την κυρία Λάτφορτ ως προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Αλβανία, διότι θυμόσαστε ότι η, όπως ίσχυσε για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο παρελθόν, θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς ειδικό για τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή αυτοί που μένουν πίσω σε σχέση με τα βιομετρικά διαβατήρια, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά στην απελευθέρωση θεωρήσεων και οι επικεφαλείς θα πρέπει να ανταμείβονται και όχι εκείνοι που παλινοδούν. Το κοσυφοπέδιο θα είναι πρόβλημα όπως είχα προβλέψει διότι δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από όλους. Η κυρία Λάτφορτ έχει δίκιο ότι αυτά που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγήσουν σε μία στρέβλωση, δηλαδή ε, όπως ίσχυσε για τους Μολδαβούς στην υπερπνηστερία που ζητούσαν ρωσικά διαβατήρια ή ρουμανικά, ε, αυτό θα ισχύσει και εδώ, δηλαδή το passport shopping, όπως λέμε. Γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελα να ψηφίσουμε ανάλογα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βάιγκλ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους εξέφρασαν ε, την υποστήριξή τους για την διαδικασία ανοίγματο όσον αφορά την ε, απαλλαγή από θεωρήσεις ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύω ότι επί της αρχής είναι λάθος να τονίζουμε τις διακριτικές γραμμές ανάμεσα στα κράτη, αλλά πρόκειται για μια απόφαση πολιτι... Ε, πρακτικής πολιτικής που ε, έχει εισάγει η Κομισιόν. Ε, μιλάμε για την αποδοχή του οδικού χάρτη και είναι σημαντικό η απελευθέρωση αυτή να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο. Πρόκειται για την ελευθερία των ανθρώπων, πολιτική ελευθερία. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Πόσελτ που το συζήτησε αυτά. Αυτό. Πριν 25-30 χρόνια την είχαμε πετύχει την ελευθερία αυτή στην πρώην Ιουκοσλαβία και είναι παράλογο τώρα να εφαρμόζουμε άλλα κριτήρια στα νέα αυτά κράτη. Στην Ευρώπη ε, έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά αστυνομικά και άλλα μέτρα. ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε μεταναστευτικά ρεύματα από τα κράτη αυτά. Για παράδειγμα, σήμερα οι δύο βοηθοί μου Ε, εξετάστηκαν προσεκτικά από τις βέλγικες αρχές, μήπως έμεναν εδώ παράνομα πριν κάποια χρόνια. Κάτι που βρίσκω απαράδεκτο και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Υπάρχουν αρκετά κανονικά μέτρα με τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε τους ε, ανθρώπους από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και από τα Δυτικά Βαλκάνια ώστε να μπορούμε να τους χορηγήσουμε ένα φυσιολογικό καθεστώς. Την αναγνώριση του Κωσόβου δεν θα πρέπει να τη συνδέουμε απαραίτητα με την διαδικασία απελευθέρωσης αποθεωρήσεις. Δεν θα πρέπει να τα θεωρήσουμε αυτά ένα ενιαίο ερώτημα. Είναι δύο διαφορετικά προβλήματα. Θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο να ασχοληθούμε με τις προϋποθέσεις πλαίσιο στο Κόσοβο με την ανάπτυξή τους ε, για μια φυσιολογική ζωή των ανθρώπων εκεί. Και φυσικά θα πρέπει να εξομαλύνουμε και τις ε, σχέσεις γειτονίας. Όσον αφορά τη Βοσνία Ζεγοβίνη, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτούς που αναφέρθηκαν στο εξής φαινόμενο. Το passport shopping, το να επιλέγει κανείς, το να ψωνίζει διαβατήρια υπηκότητες, είναι προβληματικό να το θεωρούμε αυτό φυσιολογική κατάσταση, ιδιαίτερα στις χώρες αυτές, όπου ιδιαίτερα στις χώρες αυτές που τις κυνηγάει ε, ένα ιδιαίτερο παρελθόν. Για παράδειγμα, με τις εκλογές στην Κροατία βλέπουμε ε, επανειλημμένα το φαινόμενο η ε, εκλογής από την Βοσνία να ε, αποφασίζουν το αποτέλεσμα. Δεν αναφέρεται αυτό δυνατά, αλλά πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα. Και θα μπορούσε, να, θα, θα μπορούσε να γίνει και ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό, εάν εξαπλωθεί η πρακτική αυτή. Συνοψίζοντας, η Κομισιόν βρίσκεται σε καλό δρόμο. Συμφωνώ με την απελευθέρωση αυτή. Και πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλούς συζητητές και στη δική μας Επιτροπή και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βάγκελ. Κόβατσεφ, με την εξής σύσταση για όλους να είσαστε λίγο συνοπτικοί, πιο συνοπτικοί, διότι έχω έναν μακρύ κατάλογο παρεμβάσεων και θα πρέπει να τηρήσουμε τους χρόνους εργασιών, το χρόνο εργασιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λάντφορντ. Συμφωνούμε όλοι ότι οι υπήκοοι των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που για δέκα χρόνια βρισκόταν σε μια παρόμοια κατάσταση και όταν η Βουλγαρία άρχισε τις διαπραγματεύσεις εμείς ήμασταν στη μαύρη λίστα. Εργαστήκαμε επιμακρών έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε, διασφαλίσουμε, να εγγυηθούμε μάλλον σε τέρους ότι μπορούμε και πληρούμε τους όρους και ελπίζουμε η ίδια Γενική Αρχή να ισχύσει για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα επίσης να προβώ σε ένα σχόλιο σε σχέση με την πρώην ε, ε, Δημοκρατία της Μακεδονίας Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται όχι μόνο με την προσχώρηση ή με το καθεστώς των θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι εάν η κυβέρνηση της Μακεδονίας δείξει μεγαλύτερη πολιτική θέληση, θα μπορούσε να διευθετήσει αυτά τα επιμέρους ζητήματα και αυτό δεν θα αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Εμείς λοιπόν θα υποστηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το καθεστώς των θεωρήσεων και υποστηρίζω όλα όσα προελέχθησαν. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κάτσιν. θα ήθελα να συγχαρώ την Βαρόνι Λάντφορτ για την εργασία της. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα που οφείλεται στις ε, προγενέστερες και στη σημερινή συζήτηση εδώ στην ΑΦΕΤ διότι εναρμονίζουμε τις ε, προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και για πρώτη φορά εμείς είμαστε εκείνοι που δημιουργούν τον κατάλληλο δυναμισμό. Τίποτα δεν χορηγείται δωρεάν. Η πιο σημαντική συνεισφορά σε αυτές τις ε, προτάσεις θα τη διαβάσω γιατί σας παραθέτω, είναι η αξιολόγηση της, Επιτροπής, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διενεργείται σε μηνιαία βάση που θα κοινοποιείται στο Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ενδιαφερόμενες χώρες. Αυτό χρειαζόμαστε, διότι αν μιλάμε για διακρίσεις πρέπει να είμαστε ειλικρινείς δύο χώρες, η Αλβανία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη, ε, υφίστανται διακρίσεις έναντι της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Δηλαδή, ε, είναι για δύο, πρόκειται για δύο χώρες που ε, δεν πληρούν τους όρους, τις υποχρεώσεις δηλαδή στις οποίες, ήταν, στις οποίες υπόκειντο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πιστεύω ότι ο δυναμισμός αυτός, η όθηση αυτή, οι μηνιαίες συζητήσεις στην ΑΦΕΤ και σε άλλα θεσμικά όργανα και άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεισφέρουν για μια πιο σοβαρή προσέγγιση από πλευράς ε, κυβερνητικών φορέων από την, για την, ως προς την Αλβανία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα ήθελα να σας πω ότι του χρόνου ε, μάλλον συμπληρώνονται 15 χρόνια μετά τη συμφωνία του Ντέιτον, όταν τελείωσε δηλαδή ο πόλεμος στη Βοσνία. Μετά από τις συμφωνίες του Ντέιτον. Ε, Εμείς τις επιβάλαμε και δεν μπορούν να πληρώσουν όλους τους όρους στη Βοσνία. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε αυτό το δυναμισμό και αυτές οι χώρες, αυτή η χώρα να αποδείξει την αξία της. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αντίτιμο. Ε, μόλις επέστρεψα από τη Βοσνία και το ηθικό δεν είναι ακμαίο εκεί. Νομίζω όμως ότι η σημερινή μας συζήτηση και εάν εγκρίνουμε αυτές τις τροπολογίες, τότε θα βελτιώσουμε τα πολιτικά δεδομένα στη Βοσνία και στην ευρύτερη περιοχή και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας. Από την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε για το κοσυφοπέδιο, δεν μπορούμε να, να το αγνοήσουμε. Όπως ε, ήδη ελέγχθη, η μόνη λύση μακροχρόνια για τους κοσοβάρους είναι να, να λάβουν την υπηκότητα γειτονικών χωρών. Κάτι το οποίο θα αποσταθεροποιήσει την εθνική ισορροπία σε αυτές τις χώρες και δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε για άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε, απλούστατα. Θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να, δώσουμε, να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και θαραλέοι. Διαφορετικά εμείς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που γνωρίσαμε αρκετά χρόνια πριν. Χρειάζεται λοιπόν θετική διάκριση. Αυτό χρειαζόμαστε, να δώσουμε κίνητρα σε αυτές τις χώρες, να δημιουργήσουμε επιπρόσθετη πολιτική πίεση, έτσι ώστε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και επιτεύξιμα πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενε η Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τη Βαρόνη Λάτφορντ αφενός και να πω ότι είμαι υπερήφανος ε, για τον δρόμο που διανοίγουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή ΑΦΕΤ. Κατά τις πρόσφατες εβδομάδες, σε σχέση με αυτή την κοινή πρόκληση, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για όλους και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εάν ε, ένα σώμα πρέπει να είναι υπεύθυνο, αυτό είμαστε εμείς. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα άλλα θεσμικά όργανα τι συνέβη 15 χρόνια πριν στα Δυτικά Βαλκάνια και θα πρέπει να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις και τώρα. Ευχαριστούμε κύριε Κάτσιν. Το λόγο έχει ο κύριος, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι η σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σάρα και την Τάνια για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε. Θα κοιτάξουμε την έκθεσή σου και συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επιταχύνουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων για όλες τις χώρες ε, της περιοχής με μια περιφερειακή προσέγγιση, με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και να βρούμε τρόπους για να συμπεριλάβουμε και το κοσφοπέδιο ε, σε σχέση με το ειδικό νομικό καθεστώς του. Ζητάω από την Κομισιόν να εφαρμόσει πάρα αυτά, όπως γράφει Σάρα στην τροπολογία της, ως ε, μόλις ληφθεί απόφαση το καθεστώς. Ε, εγώ ζούσα στο Σαράγεβο όταν γινόταν ο πόλεμος στην Βοσνία. Ε, και μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους ε, που τους ξέρω, για τους φίλους μου. Ε, πρόκειται για νέους ανθρώπους που αισθάνονται στη φυλακή, απομονωμένοι. Βεβαίως, οι αλβανικές αρχές, οι βοσνιακές αρχές έχουν ευθύνε. Έχουν ευθύνε να εφαρμόσουν τις προϋποθέσεις και, τους, και τα ορόσημα για όλους, ε, όπως όλοι. Ε, δεν νομίζω, Πρόεδρε, λοιπόν, ότι είναι σωστό να κρυφτούμε κάτω από το τραπέζι και να βάλουμε ένα αστερίσκο στα, στις προϋποθέσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν επί της διαφορές. Νομίζω ότι αυτό είναι απάτη. Δίνουμε ψεύτικες φρούδες ελπίδες. Ε, δημαγωγικά εντελώς βάζουμε όλους στον ίδιο κατάλογο και από δίπλα βάζουμε και ένα αστερίσκο εξαιρώντας κάποιους. Αυτό είναι απάτη. Είναι λογικό, είναι ρεαλιστικό, τους δίνουν μια προοπτική. Καλό θα ήταν, καλύτερο θα ήταν ε, να βάζουμε κάποιες ειδικέ προϋποθέσεις ε, για τις βοσνιακές αρχές. Να το αντιμετωπίσουμε σε ένα καυτό πολιτικό θέμα. Και επίση, πέρα από τι διαφορέ μεταξύ ΛΥΜΠΕ και ΑΦΕΤ, εδώ πέρα μιλάμε για τι θεωρήσει για του ανθρώπου. Αν θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, θα πρέπει να πιέσουμε τι αρχέ, να κάνουν τη δουλειά του, να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους, γιατί όπω είπατε κι εσείς, λίγη προσπάθεια να κάνουν θα τα καταφέρουν. α του βοηθήσουμε και α του υποστηρίξουμε. Α πούμε ότι είμαστε με την πλευρά του, με την πλευρά του βοσνιακού λαού. Συνεργαζόμαστε με τι βοσνιακέ αρχέ για να εφαρμόσουμε τι προποθέσει αυτέ. Α μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Είναι θέμα αξιοπιστία τη Ευρώπη. Ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία και να υιοθετήσουμε αυτό το ψήφισμα ώστε να τον πιο γρήγορα. Για το καλό του βοσνιακού λαού και για την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, Ευχαριστώ την κυρία Κοράτσα. Ο κύριος Κυρίλοφ. Και μάλιστα από αυτή τη στιγμή θα αποχωρήσω και θα αφήσω την Προεδρία στον πρώτο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Προβέρα. I think... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου έχουμε βρει ισορροπία απόψεων εδώ στην Επιτροπή. Συμφωνώ με τον ε, συνάδελφό μου κύριο Κάτσινο ότι ε, σκοπός ε, είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Την τελευταία φορά που άκουσα τον κύριο Ρέμ να μιλάει, μιλούσε για τα benchmarks αυτά και στην Βοσνία και στην Αλβανία εντός του επόμενου έτους. Όσον αφορά την όλη θέση μας, ε, πιστεύω ότι πλησιάζουμε σε μια καλή λύση, ένα θετικό πολιτικό μήνυμα προς τις χώρες αυτές, ε, με διατήρηση των γενικών αρχών μας όμως. Ε, κάτι που ε, θα επιτρέπει και θα δίνει τις άλλες χώρες να, πληρούν, να πληρώσουν τα κριτήρια. Όσον αφορά το κοσφοπέδιο, έχω δύο παρατηρήσεις όσον αφορά την παρέμβαση του συνάδελφου μου, κύριου Μπόσελτ. Να μην να μην συγχαίουμε την ε, αναγνώριση με τις θεωρήσεις. Κατά τη γνώμη μου ήταν κάπως πρώιμη η αναγνώριση, αλλά ε, δεν, ε, αυτό είναι άλλο θέμα. Άσχετα λοιπόν από τις διάφορες απόψεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, να δώσουμε προοπτική στις χώρες αυτές και όσον αφορά την πολιτική πλευρά. Η δεύτερη μου παρατήρηση, κύριε Πόσελτ, είναι ότι αναφέρατε κάποια τεράστια προβλήματα στη Μακεδονία επειδή κάποιοι ε, πολίτες έκαναν αίτηση για να αποκτήσουν ε, βουλγαρική υπηκότητα. Ε, αυτό ξεκίνησε πριν πολύ καιρό. Ε, στη 100.000 αιτήσει υπάρχουν στη Βουλγαρία, αλλά δεν έχουν λάβει υπηκότητα οι άνθρωποι αυτοί. Ε, έχει, έχουν αποκτήσει υπηκότητα μόνο όσοι κατάφεραν να αποδείξουν ότι είναι Βούλγαροι. Κάτι παρόμοιο συνέβη με τη, τους Γερμανούς στη Ρουμανία. Δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στη Μακεδονία. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό όταν συζητάμε την πολιτική της ε, παρούσας ε, κυβέρνησης ε, στην στη Μακεδονία, διότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε την πολιτική με τον εθνικισμό. Ε, είχαμε ένα παράδειγμα μιας ε, γυναίκας, ε, μιας νέας μητέρας με μωρό που, που μπήκε στη φυλακή τρεις μήνες επειδή έλαβε την υπηκότητα. Είναι ξεχωριστά θέματα αυτά. Υπάρχουν Μακεδόνες με διπλή υπηκότητα, με γερμανική υπηκότητα. Να, να μην τα συγχαίουμε τα πράγματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. La parola al collega Κύριος Κούκαν. Jedna krátka všeobecná poznámka. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία σύντομη παρατήρηση. Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι συμφωνούμε. Ότι το θέμα των θεωρήσεων για τους πολίτες ε, των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ σημαντικό. Η πολιτική κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει. Χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα, ιδιαίτερα εάν θέλουμε να δώσουμε μια σοβαρή εικόνα στους πολίτες ε, της περιφέρειας αυτής. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητη η κατάσταση εκεί. Κάποιοι από εμά ε, πιστεύουν ότι ε, γίνονται διακρίσεις, άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να περιμένουμε. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε, όμως θα πρέπει να ε, λάβουμε απόφαση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το σχέδιο της ε, κυρίας Λάτφορτ είναι πολύ καλό, είναι ρεαλιστικό, ισορροπημένο. δεν ξεχνάει ε, καμία από τις ε, ομάδες ε, της περιφέρειας αυτής και πιστεύω ότι μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε μέχρι να συμφωνήσουμε όλοι απόλυτα, διότι κάτι τέτοιο θα μας καθυστερήσει πολύ. Κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω απόλυτα το, την πρόταση της Βαρόνης Λάτφορντ. Κορνελής, τελευταίος ομιλητής. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε εκείνους που υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν ως έχει, ότι περισσότεροι μοιάζεται να λέτε ότι η πρόταση της κυρίας Λάτφορντ θέλει να δώσει με μια με το καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων σε όλες τις χώρες. Όχι, στην πραγματικότητα μία χώρα πληρεί τα κριτηρία και τέσσερις χώρες που δεν τα πληρούν. Η πρόταση της Κομισιόν αφαίρετα διαιρεί τις χώρες, τις τέσσερις υπόλοιπες χώρες, σε δύο και δύο. Ενώ η πρόταση της κυρίας Λάτφορντ διορθώνει αυτό το τεχνητό ρήγμα. Αντιμετωπίζει και τις τέσσερις χώρες που δεν πληρούν τα κριτήρια ακόμα με τον ίδιο τρόπο ότι όταν πληρώσουν τα κριτήρια θα πρέπει και οι τέσσερις μαζί να πάρουν το καθεστώς το οποίο προβλέπει απελευθέρωση από την υποχρέωση θεωρήσεων. Αυτό είναι πολύ σωστό. Επίσης αυτό που είπατε για τη μηνιαία αξιολόγηση, προκειμένου να βλέπουμε πόσο προχωρούν οι χώρες, πόσο προοδεύουν οι χώρες στην υιοθέτηση των ε, προϋποθέσεων, Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ καλή προσέγγιση, ολοκληρωμένη, για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι κάτι που χρειάζεται. Νομίζω ότι τελείωσε η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, bonjour. Καλημέρα σας. Από πλευράς Επιτροπής ε, δεν μπορώ παρά να σας υπενθυμίσω ότι λαμβάνουμε γνώση της υποστήριξής σας, της υποστήριξης αυτής της Επιτροπής ως προς αυτή την ε, πρόταση του ενδιαφέροντος ε, από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και μερικές μέρες ο Αντιπρόεδρος Μπαρό υπέβαλε στην Ολομέλεια στο Στρασβουρού εξ ονόματος της Επιτροπής τις ε, κατευθυντήριες γραμμές και την προσέγγιση της ε, Επιτροπής όταν ορίσαμε τον Ιούλιο την πρόταση σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη στην παρουσίασή μου και επίσης θα προσπαθήσω να σας υπενθυμίσω τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που ετέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής σας. Καταρχήν, σε επίπεδο επιτροπής θα ήθελα να πω ότι μέσα στα πλαίσια της κοινή πολιτικής θεωρήσεων αυτή η πρόταση τονίζει την πολιτική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων και είναι η πρώτη πρόταση που αφορά την κοινή πολιτική θεωρήσεων για μία ολόκληρη περιφέρεια. Για όλες τις χώρες αυτής της περιφέρειας σε 10 χρόνια κοινής πολιτικής για πρώτη φορά η Επιτροπή υποβάλλει μία πρόταση πολιτικής χρειάς με τεχνικά στοιχεία ως προς την προσέγγιση. Η πρώτη φορά όπου η πρόταση Επιτροπής είναι ευανάγνωστη περνώντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για να τονίσει αυτές τις προτεραιότητες που προσδίδουμε στις χώρες αυτής της περιφέρειας. Σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει μία σαφής διαδικασία. Το πρώτο στάδιο είναι η πρόταση της Επιτροπής για την απαλυφή των θεωρήσεων για, τρίτη χώρες της περιφέρειας δεσμευόμενη να συμπληρώσει την διαδικασία στο εγγύς μέλλον. Ο Αντιπρόεδρος Μπαρό ήταν ε, σαφής ως προς την ε, δέσμευση της Επιτροπής να προχωρήσει και να προτείνει του χρόνου τη συμπλήρωση αυτής της περιφερειακής προσέγγισης. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια μικρή υπενθύμηση ως προς τη προσέγγιση και τη μεθοδολογία για το θέμα της ελευθέρωσης από το καθεστώς των θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το πολιτικό πλαίσιο ήταν σαφές. Είχαμε τα συμπεράσματα της Θεσσαλονίκης που επιβεβαιώνουν την περιφερειακή προσέγγιση του καθεστώτος θεωρήσεων και που συνδέουν την άρση των θεωρήσεων με σαφείς μεταρρυθμίσεις ως προς την ελευθερία, την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Εγκρίναμε λοιπόν μία ε, κλιμακωτή προσέγγιση και θέσαμε σε εφαρμογή συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης θεωρήσεων το 2007 για πέντε χώρες της περιφέρειες έτσι ώστε να έχουμε μία εξισορροπημένη προσέγγιση για να διαχειριστούμε τον μεταναστευτικό κίνδυνο, διότι είναι ένα από τα μείζωνα κριτήρια της κοινή πολιτικής θεωρήσεων. Στη συνέχεια, για να αντιμετωπίσουμε επί, του επί της στις πολιτικές ανάγκες και να δώσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες ως προς την ε, ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις ε, μίζωνος σημασίας για την κυκλοφορία των πολιτών αυτών των χωρών. Είχαμε μια καλά διαρθρωμένη συζήτηση και έχουμε ένα λεπτομεριακό οδικό χάρτη δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες αυτού του εγχειρήματος. Πρόκειται για τεχνικές προδιαγραφές, πολύ ε, δυσχερείς αλλά αναγκαίες. Ήταν μια πολύ καλά διαρθρωμένη πρόταση και το ίδιο ισχύει και για όλες τις χώρες της περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο η οποία διαφοροποιείται ανά χώρα. Ο μείζον στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις σε όλους ε, τους τομείς ε, κλειδιά ως προς ε, θέματα ασφάλειας και χώρου δικαιοσύνης και ασφάλειας. Πρόκειται για μια διαδικασία που παρακολουθήσαμε εκ του ΣΥΝΕΝΚΙΣ το Ιανουάριο του 2008. Ξεκίνησε η διαδικασία για 1,5 χρόνο. Παρακολουθήσαμε τις μεταρρυθμίσεις όλων των χωρών της περιφέρειας. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες επικυρώθηκαν από εκθέσεις μας που βασίζονται όχι μόνο σε πληροφορίες επί χάρτου, αλλά μετά από αποστολές με εθνικούς εμπειρογνώμονες. Συμμετείχαν δηλαδή και οι εθνικοί εμπειρογνώμονες, κάναμε αποστολές αξιολόγησης και είδαμε κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις ισχύουν in situ. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί στο Δινεκές από πλευράς ε, Επιτροπής. Πώς ορίσαμε τον κατάλογο αυτό. Κάναμε μία αυθαίρετη επιλογή όταν προτείναμε τις τρεις χώρες. Νομίζω ότι η Επιτροπή κατάρτισε λεπτομεριακές εκθέσεις με βάση την πρόοδο που είχε επιτελεστεί από τις πέντε χώρες. Η αξιολόγηση της Επιτροπής ε, την αξιολόγηση την συμμερίστηκαν όλα τα κράτη στο Συμβούλιο και συζητήθηκε και με τις χώρες της ε, περιφέρειας. Η πρότασή μας επιβεβαιώνει ότι όλα τα κριτήρια που ορίζονται στον οδικό ε, χάρτη πληρούνται για τη Σερβία και το Μαυρο... Μαυροβούνιο δεν προβήκαμε σε μία αυθαίρετη αξιολόγηση. Θεωρήσαμε ότι υπάρχει μία δυναμική συνέργεια για αυτές τις δύο χώρες. Και όταν καταρτήσαμε την πρότασή μας, όλα είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Απλώς έπρεπε να ε, πληρωθούν και ορισμένα άλλα μέτρα που είδαμε από αυτές τις χώρες, όπως είχαν οριστεί επί χάρτου. Και προβλέπουμε κατά τα μέσα Οκτωβρίου να προβούμε σε αποστολές αξιολόγηση που θα ορίσουν κατά πόσο πληρούνται όλα τα κριτήρια, τα κριτήρια του οδικού χάρτη. Σε αυτά τα πλαίσια θεωρήσαμε ότι η Αλβανία και η Βοσνία έχουν επιτελέσει μεγάλη πρόοδο στα πλαίσια των συζητήσεων ως προς την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, αλλά για τα τέσσερα μεγάλα μπλοκ κριτηρίων θα πρέπει να προβλέψουμε συγκεκριμένες δράσεις και μετά να επαληθεύσουμε την εφαρμογή τους έτσι ώστε να συμπληρώσουμε τα κριτήρια τα οποία ορίζονται. Βεβαίως μπορούμε να λάβουμε μια πολιτική απόφαση και να πούμε ότι αυτά που πληρούνται αρκούν. Ακόμα και αν έχουμε ορίσει λεπτομεριακά κριτήρια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις αυτών των ε, αποφάσεων για το μέλλον, για την κοινή μας πολιτική θεωρήσεων και για την αξιολόγηση αυτή της Κομισιόν αποκοινούμε εσάς, τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη για την κοινή πολιτική θεωρήσεων. Δηλαδή, κατά πόσο η πίκο ενός κράτους μέλους υπόκεινται σε καθεστώς θεωρήσεων ή έρονται αυτά τα κριτήρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι τίθενται σε εφαρμογή αυτά τα κριτήρια, έχουμε επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και η πείρα μας στα Βαλκάνια το αποδεικνύει αυτό, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο θέλουμε να προβούμε σε μία αξιολόγηση η οποία να είναι λεπτομεριακή, κρατώντας όλους τους πολιτικούς στόχους. Και η πρόταση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει αυτά τα κριτήρια, αυτή την εξισορροπημένη προσέγγιση για να προχωρήσουμε περαιτέρω και να συμπληρώσουμε την ε, διαδικασία με μια νέα πρόταση τη στιγμή που τα κριτήρια θα πληρούνται από όλες τις ε, χώρες της περιφέρειας. Θα ήθελα επίσης ε, να σχολιάσω το εξής. Διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του Κοινοβουλίου που επιβεβαιώνει τη σημασία αυτού του ζητήματος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε την πολιτική υποστήριξη του Κοινοβουλίου στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματο. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι ήδη έχουμε την πείρα την εμπειρία των αστερίσκων, όπως στη Ρουμανία, ίσχυσε στη Ρουμανία το 2001 και στα πλαίσια αυτής της εμπειρίας τότε συντάχθηκε μία έκθεση Επιτροπής που δεν ήταν τόσο λεπτομεριακή όπως το τωρινό εγχείρημά μας και η έκθεση αυτή δεν δημοσιεύθηκε. Με βάση όμως αυτή την έκθεση το Συμβούλιο, το ίδιο το Συμβούλιο αποφάσισε να διαγράψει αυτό τον αστερίσκο και να διαγράψει την υποχρέωση θεωρήσεων για τους Ρουμάνους υπηκόους. Η έκθεση του Κοινοβουλίου για αυτή, σε αυτή την έκθεση δεν ακολουθεί αυτή την προσέγγιση, αυτό το νομικό πλαίσιο. Τώρα, εν συντομία, θα απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που ετέθησαν από μέλη ως προς τον έλεγχο της όμορης περιοχής μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Αναφέρθηκε στην πρώτη της Επιτροπής η ε, Επιτροπή θα κάνει αποστολές in situ και θα δει κατά πόσο αυτό το working arrangement ισχύει που υπεγράφει μεταξύ Ulex και σερβικών αρχών και στα μέσα Οκτωβρίου θα συντάξουμε έκθεση για να δούμε και να επαληθεύσουμε κατά πόσο ισχύει το επίπεδο ασφάλειας για κάθε διέλευση των συνόρων και οι ίδιες προδιαγραφές και για αυτή την περιφέρεια. Οι προδιαγραφές είναι οι ίδιες, οι ανάγκες ασφάλειας είναι επακριβώς οι ίδιες και υπάρχει και η ίδια προσέγγιση. Τώρα, για το θέμα των μικροχωρών, τα μικροετά και την άρση των θεωρήσεων, όπως, όπως θα συζητήσουμε το απόγευμα στη ΛΥΜΠΕ. Η Επιτροπή ήδη το 2006 αξιολόγησε και ανέφερε ότι αυτές οι χώρες μπορούν να περάσουν στη θετική λίστα. Αλλά επειδή υπάρχει αυτός ο νομικός σύνδεσμος και για να εγγυηθούμε μία αμοιβαιότητα κατά 100% σε σχέση με τους δικούς μας υπηκόους, δηλαδή για όλους τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρήσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε κοινοτικέ συμφωνίες άρσης ε, θεωρήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική πλαισίωση από ό,τι ισχύει στα Δυτικά Βαλκάνια και θεωρούμε ότι ο σύνδεσμος αυτός, η γενικότερη διαδικασία είναι διαφορετική, διότι για αυτές τις χώρες υπάρχει επιβεβαίωση ευρωπαϊκής συμμετοχής, δηλαδή προσχώρησης, έχει επιβεβαιωθεί σε πολιτικό επίπεδο πολλές φορές και έτσι η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν, χρειάζεται, δεν χρειάζονται αυτές οι συμφωνίες. Μετά από τη δημοσίευση και την εφαρμογή αυτής της πρότασης. Άρα η πλαισίωση είναι διαφορετική. Οι σχέσεις που έχουμε με τα Δυτικά Βαλκάνια και η διαδικασία προσχώρησης, δηλαδή η ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των χωρών, μας οδηγεί στο να προωθήσουμε μία διαφορετική διαχείριση του καθεστώτος ως προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων σε σχέση με την προσέγγιση που είχαμε για αυτά τα μικροκράτη, μικροετά. Το τελευταίο σχόλιο αφορά το δικό σας ε, σχολιασμό, πολλών μελών τι λένε, ως προς το passport shopping. Είναι κάτι το οποίο μας ε, απασχόλησε επί μακρόν όταν ορίσαμε τον οδικό χάρτη και την όλη διαδικασία. Ζητήσαμε από τις ενδιαφέρομενες χώρες ε, πληροφορίες και εγγυήσεις σε σχέση με το χρόνο για την χορήγηση διαβατηρίων, δηλαδή με βάση συγκεκριμένες υπηκότητες. Έχουμε στατιστικά δεδομένα από, τρίτες χώρες, όπου, από τρεις χώρες όπου προτείναμε την απελευθέρωση. Έχουμε λεπτομεριακές εκθέσεις, δηλαδή πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει χορήγηση υπηκότητας από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική απόφαση για την απόκτηση υπηκότητας και πόσο καιρό χρειάζεται για την χορήγηση διαβατηρίου. Εάν, όπως είπε ο πρόεδρος Μπαρό, ολοκληρώσουμε τη διαδικασία το 2010 με μία πρόταση τη στιγμή που πληρούνται όλα τα κριτήρια, τότε νομίζω ότι δεν θα διατρέχουμε κίνδυνο για passport shopping. Ο κίνδυνος θα είναι αρκετά περιορισμένος. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η εισηγήτρια για να μας ε, μιλήσει για τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ, πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές που ήταν και η πλειοψηφία που συμφωνούν με τη βασική κατεύθυνση της νομοδότησής μου, που όπως είπα ευθυγραμμίζεται γενικά με το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Φεϊόν από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Στις δύο αυτές επιτροπές προτείνεται πιστεύω, μια ισορροπημένη προσέγγιση, όπως ε, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Είναι πολιτική, διότι ε, περιλαμβάνει και τις πέντε χώρες ε, της περιφέρειας. Εξαλείφει δηλαδή τις αμφιβολίες σχετικά με την πολιτική βούληση όσον αφορά τις πέντε αυτές χώρες, αλλά αλλά διατηρείται η ε, απέτηση για πλήρωση των benchmarks. Ε, λυπάμαι που έφυγε ο Δ. Τάνοκ, ε, ε, διότι διαφωνώ μαζί του. Βέβαια, είμαι υποχρεωμένη να διαφωνήσω μαζί του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, λέει εδώ πέρα και συμφωνώ με αυτό ότι ότι δεν θα πρέπει οι, οι χώρες που ηγούνται να καθυστερήσουν λόγω της καθυστέρησης των άλλων, ε, εφόσον δηλαδή πληρούν τα κριτήρια. Η γνωμοδότηση και η έκθεση αυτή ενοποιεί το πολιτικό μήνυμα, αλλά διατηρεί την τεχνική προσέγγιση και δεν υποσκάπτει την όλη διαδικασία του οδικού χάρτη. η αίσθηση ιδιοκτησία και η εξουσία παραμένουν στα χέρια της Επιτροπής. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπής όταν... όταν λέει ότι δεν υιοθετούνται εδώ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Ρουμανία του 2001. Λέει ότι οι πιο αργές ε, χώρες θα ε, είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούν τα κριτήρια. Κύριε Πρόεδρε, Διαφωνώ μαζί σας. Όταν είπατε ότι προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απεβολεί τα προνόμια του. Έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά αναδομούμε την πρόταση ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή να μην έχουμε δύο προτάσεις. Ελπίζω να είναι σαφές αυτό. Συμφωνώ και επικροτώ με τις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Πόσελτ, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ορισμό της ασφάλειας με ευρύ στρατηγικό τρόπο. Ε, συμμετείχα στη ΛΥΜΠΕ, δεν υπάρχει κανένας που να ενδιαφέρεται περισσότερο από μένα ε, για την για την ενότητα στη διαδικασία για τις θεωρήσεις, αλλά οι χώρες αυτές υπόκεινται σε benchmarks τα οποία είναι πολύ πιο ευρεία από, τα από το θέμα των ταξιδιωτικών εγγράφων. Εάν υποσκάψουμε τη σταθερότητα στις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων, ε, ε, θα οδηγηθούμε σε έλλειψη σταθερότητας. μειοψηφία των ομιλητών τη επιτροπή μα διαφώνησαν με την έκθεση αυτή και νομίζω ότι αυτό κυρίω είχε να κάνει με το θέμα του κοσφοπεδίου. Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να υποσκάψουμε τη θέση των ε, κρατών μελών που δεν έχουν ε, αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παντρέψουμε την ε, διπλωματική και νομική αυτή θέση με τη δυνατότητα να είμαστε ρεαλιστικοί όσον αφορά την πρόοδο στο θέμα του κοσφοπεδίου. Υπάρχει μια διαφορά στην διατύπωση ανάμεσα στην γνωμοδότησή μου και την έκθεση της κυρίας Φαγιών. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ έγραψα τη γνωμοδότησή μου πριν ε, οριστικοποιήσει η κυρία Φαγιών την έκθεσή της, ε, αλλά ουσιαστικά μεταδίδουμε το ίδιο μήνυμα. Δεν νομίζω ότι έχω πολλά άλλα να πω. Να συμφωνήσω όμως με την κυρία Κορνέλησεν ότι όσα προτείνονται εδώ στόχο έχουν την ίση μεταχείριση των τεσσάρων χωρών που δεν είναι ακόμα επιλέξιμες. Η δυσκολία στην πρόταση της Επιτροπής είναι ότι προτείνουμε να συμπεριληφθούν στον κανονισμό αυτόν όλε οι χώρε ε, που ήταν επιλέξιμε μέχρι την 1η Ιουλίου. Αλλά αν το κάναμε αυτό θα ήταν δύσκολο να συμπεριλάβουμε τι δύο τελευταίες χώρες. Ε, ήδη ήταν μια ε, πρόταση σε δύο δέσμες. Το να το κάνουμε αυτό λοιπόν πρόταση τριών δεσμών δεν είναι τελείω περίεργο. Κλείνοντα, επικροτώ την ευρία υποστήριξη της Επιτροπής. Ελπίζω αυτοί που δεν συμφωνούν να δεχτούν τη ρεαλιστική προσέγγιση για το Κόσοβα. Όσοι πιστεύουν ότι υπονομεύω τα, την προσέγγιση των benchmarks, ελπίζω να δεχτούν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ε, απαλλάσσουμε από θεωρήσεις εάν δεν πληρωθούν τα benchmarks και για το δικό τους καλό και για τη δική μας την ασφάλεια. Ελπίζω η Επιτροπή να μπορέσει να ε, υποστηρίξει την έκθεση στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ε, e ευχαριστώ για τη δουλειά σας και για τον ενθουσιασμό σας. Και υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι η τελική προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι η 1η Οκτωβρίου και οι τροπολογίες θα παρουσιαστούν στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Πάμε στο προηγούμενο σημείο. Σας ζητώ μία-δύο, ένα-δύο λεφτά ε, υπομονής στο μέσο για τη σταθερότητα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Μπράντνερ, για να αναδιατυπώσει τη διατύπωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ευχαριστώ που μου, ζητά, που μου δίνει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που επανέρχομαι. Ε, ευχαριστώ που έχετε την υπομονή να κάτσετε τόσο αργά. Δύο-τρία λεφτά χρειάζομαι υπομονής γιατί αξίζει προσοχή σε αυτό το σημείο. Ε, υποστηρίζουμε και συμφωνούμε με την απόφαση του ΔΕΚ και με την προσέγγισή σας να επεκτείνετε τις προμήθειες και να τις ανοίξετε παγκοσμίω. Δεν είμαστε ενάντια στην αύξηση του 10% ε, στο άρθρο 4.1, όμως θα θέλαμε μια καθαρότερη εικόνα της στρατηγικής και του στόχου και να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι στιγμής πριν υπάρξει επέκταση. Επίσης θα θέλαμε να ενημερωθούμε περισσότερο για το Κέντρο Αντιτρομοκρατίας στο Αλγέρι. Γενικώ πώς θα ήθελα να πω ότι θα θέλαμε να υπάρχουν πιο ε, επιμελείς εκθέσεις και λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε για τα πρώτα στάδια της όλης διαδικασίας που είδαμε. Και το τελευταίο σημείο, τι γίνεται με την ε, οικοδόμηση ε, εταιρική σχέσης για την ειρήνη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει διασκέψεις, εργαστήρια κτλ. Νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα θέλαμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επίσης, μίλησαμε για τα προβλήματα ε, της ε, χρηματοδότησης ε, που έχουν πάει ε, στο μέσο για τα τρόφιμα. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούβης Καλαβέρα. Ευχαριστώ τους βουλευτές, την κυρία Μπράντνερ και την Επιτροπή ΑΦΕΤ για τη σημαντική υποστήριξη που μας δίνει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του μέσου σταθερότητας τα τελευταία τρία χρόνια από τη στιγμή που δημιουργήθηκε από το 2007 μέχρι σήμερα και για τη θετική ανάλυση της εισηγήτριας σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λόγους που την οδήγησαν στην τροπολογία της νομικής βάσης, όπως την υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Επίσης, θα θέλαμε να δοθούν οποιασδήποτε διευκρινήσεις θέλετε, εσείς ως ΑΦΕΤ, για να μην έχετε την αίσθηση ότι δεν έχετε αρκετές πληροφορίες ό,τι αφορά τη στρατηγική και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ε, υπό το άρθρο 4.1. Θα καταλαβούμε καλύτερα τις ανάγκες σας, γιατί πιστεύουμε ότι αν αυξήσουμε τα ποσοστά από το 7% στο 10%, αυτού του πολύ σημαντικού άρθρου, που αφορούν ε, την ασφάλεια των ατόμων, ε, την κρίσιμη υποδομή, τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους πολίτες και χρειαζόμαστε ουσιαστικά κονδύλια για να αναπτύξουμε στρατηγικές πιο φιλόδοξες. Γιατί η διασυνοριακή και κίνδυνοι όπως οι πανδημίες, οι μεγάλες επιδημίες, οι μεγάλες υποδομές, παροχή ενέργειας κτλ. δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με λίγα κονδύλια ή καταπολέμηση ας πούμε της εγκληματικότητας. Επομένως η αύξηση της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντική για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτές τις απειλές. Επίσης, Οποιαδήποτε συνεργασία και διάλογο θέλετε να έχουμε, είμαστε διατεθειμένοι να σας το εξασφαλίσουμε. Εμείς κάναμε μία προσπάθεια στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του IFS. Ε, προσθέσαμε ένα παράρτημα με, μονομένα δελτία για το κάθε πρόγραμμα όπου παρουσιάζουμε όλες τις δυσκολίες που ε, έχουμε. Ούτω ή άλλω τα προγράμματα αυτά δεν είναι παραδοσιακά. Μιλάμε για περιοχέ που βρίσκονται σε κρίση και τα κριτήρια φυσικά είναι διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων για την ειρήνη, έχουμε να γνωρίσει τι ε, δυσκολίε για να εφαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα και για να έρθουμε σε επαφή με πιο διαφορετικό τρόπο με την κοινωνία των πολιτών. Ε, δύο πράγματα ήταν σημαντικά φέτος. Ήταν περισσότερο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και έχουμε και παραγγείλει μία μελέτη όπου οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όσοι γνωρίζουν Και όσοι γνωρίζουν την ε, δομή της ε, Κομισιόν θα ξέρουν ότι για να εφαρμόσουμε το 4-3 θα πρέπει να σεβαστούμε τις πολύ αυστηρές δημοσιονομικές προϋποθέσεις. Έχουμε λάβει μία έκθεση με συστάσεις, θα σας τη δώσουμε, θα τη δώσουμε στην εισηγήτρια και θα εξετάσουμε την έκθεση αυτή για να ε, οργανωθούμε, να οργανώσουμε τις επαφές μας ε, με την κοινωνία των πολιτών. Τελευταίο, καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες της ΑΦΕΤ σε ό,τι αφορά τις περικοπές στη γραμμή του, προ... του προϋπολογισμού. Και καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να το θέσετε αυτό στην Επιτροπή Προπολογισμών, ούτω ώστε να δοθεί ιδέουσα προσοχή από τις αρχές. Δεν θέλω να σας κλέψω περισσότερο χρόνο. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες. Στρέφομαι και προς τους συναδέλφους του Συμβουλίου. Το θέμα και σας ε, διαβεβαιώνω ότι το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι τις ανάγκες αυτής της πρότασης ε, για να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση, γιατί το μέσο σταθερότητας θα πρέπει να δώσει μια συνολική απάντηση στους κινδύνους ε, αστάθειας, να δώσει απαντήσεις σωστές σε θέματα ασφάλειας κτλ. Αυτά κλείνουν εδώ οι εργασίες μας και θα ξαναπούμε το απόγευμα.